Hello everyone. Γεια σας, παρακαλώ καθίστε και ετοιμάσετε τις κάρτες σας για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την σημερινή μας ψηφοφορία. Έτοιμοι όλοι. Η πρώτη έκθεση είναι η εφαρμογή των μέσων παρέχει η ΚΑΠ στους γεωργούς μετά τη μεταρρύθμιση του 2013. Αρχίζουμε με τη συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά ελέγχουμε τη 13 αρχίζει η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται 14 υπέρ. Κατά αποχές απο... Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη, 15 υπέρ. Κατά αποχές ας ελέγξουμε, μάλλον 15 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε, ελέγχουμε τώρα. Λυπάμαι, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο.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 αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ. Κατά, αποχές Ελέγχουμε την 63 ηλεκτρονικά. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 75 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 σε δύο τμήματα. Πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 80 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά η οποία και άρχεται. Και πέρας. Και εγκρίνεται. Τώρα ψηφίζουμε την ερμηνεία και εφαρμογή της Διοργανικής Συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ένα Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρία Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πέντε Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έξι Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά ελέγχουμε την 10 άρχεται η ψηφοφορία πέρας Ισοψηφία, άρα απορρίπτεται. 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ας ξαναψηφίσουμε γιατί δεν είμαι σίγουρη. 11 υπέρ. Κατά. Ε, θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 11. Πέρας. Εγκρίνεται. 12. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε τη 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε την 14. Ε, Με συγχωρείτε, ε, ψηφίστε διαφορετικά από το ένα θέμα στο άλλο πολλές φορές, πέρας, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ, κατά αποχές ελέγχουμε την 31 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 32 υπέρ. Υπάρχει κάτι το οποίο μπορείτε να μοιραστείτε μαζί μας, γιατί επικρατεί θυμηδία και θα ήθελα να ξέρω γιατί. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 35 άρχεται ψυχοφορία. ψηφοφορία και πέρας και απορρίπτεται και εγκρίνεται και εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά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 και πέρας και εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην επόμενη. Next. Η επόμενη έκθεση. Επιφυλακτικότητα προς τον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη. Αρχίζουμε την τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Το δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά απορρίπτεται. Όχι. Ας κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση στην 42. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται η 42. 43.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 αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση στην 88 αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται απορρίπτεται. 96 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, ε, απορρίπτεται συγγνώμη, η 2 εγκρίνεται, η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 3 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 3. Αρχίζει η ψηφοφορία. Κυρία Ντολέ, έχετε την κάρτα σας. Λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 38 το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία του σχεδίου ψηφίσματος, έτσι όπως τροποποιήθηκε, αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαφανής και υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων στις Συγγνώμη, βιώσιμο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τομέα ιδιωτικού 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Δεν είστε πολύ ενεργοί βλέπω. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 15 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά Δεκαοκτώ. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 21 το πρώτο μέρος υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πού βρισκόμαστε, λέει η πρόεδρος. Θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση στην 23. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση του, ε, του πρώτου μέρους της τροπολογίας 31. Αρχίζει η ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος της 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 32. Αρχίζει η ψηφοφορία. αν δεν μας πείτε πώς ψηφίζετε, δεν ξαναπροχωρώ σε αυτό το παιχνίδι. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 33. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Το πρώτο μέρος. Το δεύτερο. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 34. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 35. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 30, ε, εγκρίνεται, συγγνώμη, 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 35 υπέρ κατά αποχές Οι σοσιαλιστές είστε υπέρ ή κατά. Λοιπόν, Α επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. απόχέ Εγκρίνεται. 54 υπέρ, δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 56. Υπέρ. 56 κατά αποχές. Κανένας δεν υπερψήφισε αυτή την τροπολογία. Απορρίπτεται. 57. Υπέρ. Κατά αποχές. Είστε πάρα πολύ γρήγοροι κυρία Πρόεδρε. Έγινε λοιπόν κάποια σύγχυση με το 54, το πρώτο δεύτερο μέρος, το 56 δεν ξέρουμε τι έγινε, θα μπορούσαμε να επανέλθουμε στην 56. Λοιπόν, ε, πάμε στο δεύτερο μέρος 54. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 57. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 58. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 59. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 60. Πρώτο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 61. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 62. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63, υπέρ, κατά. Α, καταπίπτει 63. 66, υπέρ, κατά, αποχές. Επαναλαμβάνουμε, 66, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 75, υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 το πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82. Υπέρ, κατά, αποχές. 82 επαναλαμβάνει η πρόεδρος. Υπέρ, κατά, αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 82. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 84 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται 87 υπέρ κατά, απόχέ εγκρίνεται. 88 υπέρ, κατά, Αποχέ απορρίπτεται. 89 υπέρ, κατά, Αποχέ απορρίπτεται. 90 υπέρ, κατά, Αποχέ απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, απόχέ. Ηλεκτρονική επαλήθευση 91 αρχίζει ψηφοφορία. Λίγη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 95. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 96. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 97 απορρίπτεται 98 υπέρ κατά ε, απορρίπτεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά ε, αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε το σχέδιο, νομοθετη... το... σχέδιο ψηφίσματος στο σύνολό του Λίγη ψηφοφορία, λίγη ψηφοφορία εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις. Τα αποτελέσματα της προηγούμενης ψηφοφορίας 61 προς 1. Δεν εμφανίστηκε στην οθόνη. 61 υπέρ, ένας κατά και καμία αποχή, λέει πρόεδρος, για την ε, προηγούμενη έκθεση. Ψηφίζουμε τη δέσμη μέτρων στρατηγικής για τις δημόσιες συμβάσεις. Τροπολογία 7, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8, υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος για την 8, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίθηκε. Εννέα. υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Ή εγκρίθηκε. Ας ελέγξουμε και την εννέα, παρακαλώ. Σας ζητώ συγγνώμη. Αλλά άμα δεν σηκώνετε καλά τα χέρια σας δεν βλέπω. Πέρας και εγκρίθηκε.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 στην ημερήσια τέταξη. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία.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 So, colleagues, I would like to encourage... Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν στην συζήτηση για την επόμενη ανταλλαγή απόψεων, σας παρακαλώ, βγείτε από την αίθουσα, γιατί θα συνεχίσουμε κατευθείαν. Σας ευχαριστώ και να περάσουμε λίγο λοιπόν στο 13 της της διάταξης. Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Έχουμε να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ. Να συνεχίσουμε με το 13 λοιπόν τη ημερήσια έταξη. συνταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με το γενετικό κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα δώσω παρά αυτά το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας καλέσατε να παρουσιάσουμε την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά την παραποίηση φαρμάκων. Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 118 της σχετικής οδηγίας, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προβλέπουν αποτελεσματικές και αναλογικές κυρώσεις για να αποφεύγουν τέτοιες παραποίησεις φαρμάκων σε ό,τι αφορά και τα έκδοχα σε ό,τι αφορά και τι δραστικέ ουσίε. Θα πρέπει λοιπόν τα κρατημέλη να κοινοποιούν τα μέτρα αυτά προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 118α ε, ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προδιαγράφει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι αφορά τα μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη-μέλη και την αποτελεσματικότητά τους. Η έκθεση λοιπόν αυτή εγκρίθηκε 26 Ιανουαρίου του 2018. Έγινε εξωτερική ανάθεση μιας έρευνας και μελέτης, η οποία μας βοήθησε για την εξαγωγή της έρευνας και πλέον και η μελέτη μας από την έκθεση είναι στο διαδικτύο δημοσιευμένη. Τα απορίσματα λοιπόν σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, τα κατημέλη και τις κυρώσεις. Να έχουμε υπόψη μας καταρχάς ότι μιλάμε για παραποιημένα φάρμακα. Εξορισμού λοιπόν είναι δύσκολο να αξιολογηθεί, να εκτιμηθεί αυτός ο κλάδος, αυτός ο τομέας. Οι σωματικές βλάβες, ε, καλύπτονται να έχουμε υπόψη μα από το ποινικό δίκαιο σε όλα τα κρατη και τα κράτη-μέλη επίση επιβάλλουν διοικητικέ κυρώσει για παράνομη χρήση φαρμάκων. Αυτέ οι κυρώσει λοιπόν στα κράτη-μέλη συμπληρώνονται και από συγκεκριμένε κυρώσει για την παραποίηση φαρμάκων, εκδόχων, ταστικών ουσιών όπω προβλέπεται στο 118α. 26 λοιπόν έχουν εισαγάγει αλλαγέ στην νομοθεσία τους για να εφαρμόσουν το 118α και ένα κράτο μέλος ε, άλλαξε και το ποινικό του κώδικα για να ανταποκριθεί στις ε, προδιαγραφές ε, του Ιατρικού Συμβουλίου και ένα κράτο μέλο δεν άλλαξε την νομοθεσία του γιατί είχε την αίσθηση ότι ήδη υπήρχαν σχετικέ κυρώσει και πριν την εφαρμογή του 18α. Άρα, οι τρέχουσε κυρώσει για την ε, παραποίηση των φαρμάκων εκδόχων δαστικών ουσιών είναι πρόστιμα, φυλάκιση και διοικητικά μέσα, όπω, για παράδειγμα απόσυρση προϊόντων, απόσυρση αδειών κτλ. Σε όλα τα κράτη-μέλη, κάποιε από τι δραστηριότητε αυτέ είναι ποινικού δικαίου και σε 21 κράτη-μέλη η παραγωγή, εξαγωγή, εισαγωγή, διανομή τέτοιων φαρμάκων συνεπάγονται ποινικέ κυρώσει και σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε αστικές κυρώσεις και όχι ποινικέ όπως πρόστιμα. Υπάρχει μέγιστη περίοδος φυλάκισης από 1 έως 15 χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την παραποίηση φαρμάκων. Όλα τα κρατημέλη μελη επίσης εφαρμόζουν ποινικέ και αστικές κυρώσεις και πρόστιμα 4.000 στη Λουθιανία έως 1 εκατομμύριο στην Ισπανία. Και για Έχουμε 23 κράτη-μέλη που εφαρμόζουν ε, ποινικέ ε, ε, κυρώσει για παραβίαση φαρμάκων, 14 σε ό,τι αφορά τα έκδοχα. Σε ό,τι αφορά τι αστικέ ουσίε, 26 κράτη-μέλη εφαρμόζουν ποινικά ή αστικέ κυρώσει και για τα έκδοχα 20 κράτη-μέλη. Επίσης, να σημειώσουμε ότι όλα εκτό από τρία τα κράτη-μέλη έχουν εισαγάγει επιπρόσθετες διοικητικές κυρώσει για την παραποίηση φαρμάκων, εκδοχών και δραστικών ουσιών. Αν δούμε λοιπόν τώρα την αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών που ακολουθεί. Όπω σα είπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να προσμετρηθούν όλα αυτά. Γιατί εγγενώ είναι παράνομε οι δραστηριότητε αυτέ. Και επίση αυτό αποτέλεσε μία από τι δυσκολίε που αντιμετώπισε ε, η εταιρεία στην οποία αναθέσαμε τη μελίτη γιατί προφανώ πρέπει να συλλέξει όλα αυτά τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, τη. Ε, και Αλλά σε γενικές γραμμές ε, ε, για να υπάρχει σωστή αποτελεσματικότητα και να αποτρέπεται αποτελεσματικά η πώληση των παρανομαφαρμάκων θα πρέπει να υπάρχει συνδυασμό και ποινικών και αστικών κυρώσεων. Ενδεχομένω να χρειάζονται και να αποδεχθεί η συγκεκριμένη βλάβη που έχει προκληθεί από το φάρμακο. Αυτό ισχύει για τα πιο πολλά κράτη-μέλη. Ε, ένα άλλο στοιχείο. Η μέγιστη περίοδο φυλάκισης τριών ετών ως ε, προδιαγραφή μπορεί να διευκολύνει την ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη και ένταλμα για την ενέργεια ερευνών. Και έτσι λοιπόν, ε, συμπερασματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι έχει εφαρμοστεί το έργο α με αποτελεσματικό και σωστό τρόπο. Θα μπορούσαν τα κράτη-μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολή ποινικών κυρώσεων ή διοικητικών κυρώσεων σε ό,τι αφορά τα φάρμακα, δραστικέ ουσίε και έκδοχα. Και επίση χρήσιμο θα ήταν να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν επαρκή πόροι και ανθρώπινη πόροι, προσωπικό, για να γίνουν όλα αυτά μέσω εκπαίδευση κατάρτιση νέων με υπαλλήλων και η καλύτερη καταμέτρηση και διανομή των δεδομένων θα μπορούσε να βοηθήσει καλύτερα προκειμένου να ξέρουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων γιατί είναι πολύ δύσκολο να έχουμε σωστά και απακριβή στοιχεία σε ό,τι αφορά την έκταση της παραποίησης στην ευρωπαϊκή αγορά. Και τέλος, ε, χρειάζονται μέτρα αποτροπής, κυρώσεις ε, οι οποίες θα δρουν αποτρεπτικά. Αυτό θα είναι δυνατόν μόνο με τη σωστή συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων των πρακτικών σε ό,τι αφορά την των γνωμοθεσία. Εδώ συνεργαζόμαστε πολύ στενά με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κροστέτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και να ευχαριστήσω την Επιτροπή για τις εξηγήσεις που μας έδωσε, διότι αυτό το άρθρο 178α για τα παραχαραγμένα φάρμακα θα πρέπει να μεταφερθεί σωστά. Τα συμπεράσματα είναι θετικά, αλλά η παραποίηση φαρμάκων είναι ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό για εμάς γιατί αυτή η παραχάραξη μπορεί να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες. Είναι ένα σοβαρό θέμα δημόσιας υγείας. Μιλάμε για την εφοδιαστική αλυσίδα παράνομων φαρμάκων και την επιγραμμική αγορά τους, παράνομη αγορά. Και πέρα από τις κυρώσεις στις οποίες αναφερθήκαμε, μας ενδιαφέρει ο ρόλος το, του αντικτύπου της επιγραμμικής πώλησης παραχαραγμένων φαρμάκων. Η Επιτροπή βρήκε ένα συσχετισμό μεταξύ του ανοίγματο επιγραμμικής πώλησης και της παραχάραξης αυτής ή υπάρχει συσχετισμός μεταξύ επιγραμμικής ε, πώλησης και σκευασμάτων και τέτοιων σκευασμάτων ε, είναι ένα προτιμησιακό κανάλι πωλήσεων. Και πριν από τις κυρώσεις η Επιτροπή γνωρίζει κατά πόσο είναι αποτελεσματική η έλεγχη για τις επιγραμμικές πωλήσει. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάουκεν. Χάουκεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε πράγματι συζητήσει αυτά τα θέματα και δεν μας ενδιαφέρει μόνο να δούμε κατά πόσο υπάρχουν ποινικέ κυρώσεις, σίγουρα υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ορίσουμε αυτό το φαινόμενο καλύτερα και να το οριοθετήσουμε, γιατί για αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει απλώς να υπάρχει σωστή σήμανση, αλλά και ανιχνευσιμότητά τους για να ξέρουμε από πού προέρχονται. Για διαφορετικά ε, ίσως συνεχίσουν να υπάρχουν καταχρήσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε περισσότερες προδιαγραφές για την ανιχνευσιμότητά τους. Και θα πρέπει να προβλέψουμε και ποινικέ κυρώσεις, γιατί είναι αξιόπινες πράξεις. Και δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδιάφοροι απέναντι σε ένα τέτοιο ε, φαινόμενο. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, αναχαιτιστικά μέτρα. Μην ξεχνάμε πόσα χρήματα βρίσκονται επιτάπητος ή διακυβεύονται. Ο κύριος Λίζε. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκθεση αυτή. Αλλά θα ήθελα να επιμείνω λίγο, γιατί η έκθεση ήταν πάρα πολύ επίσημη. Τι έκαναν τα κράτη-μέλη, πολύ τυπική. Τι νομοθεσίε τροποποιήθηκαν και το καθεξή. Εμεί αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να λυθεί το πρόβλημα. Μια εκτίμηση λοιπόν θα ήθελα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έγινε πρόοδο σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των παραποιημένων φαρμάκων. Και να επαναλάβω επίση από την ερώτηση που έθεσε και η Φρανσουά Γκροστέτ. Είχαμε πληροφορίε ότι στο διαδίκτυο ιδιαίτερα είναι πολύ δεδομένη η παραποίηση φαρμάκων. Ε, βάλαμε λοιπόν το σύστημα αυτό με τη σφραγίδα. Ε, πόσο έχει βοηθήσει, πόσο έχει προχωρήσει το σύστημα αυτό, μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώ πώς εκτιμά την κατάσταση, υπήρξε κάποιο αντίκτυπο, περιορίστηκε το πρόβλημα, Πώ πήγαν τα πράγματα, γιατί με αυτό που μα ενδιαφέρει είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Και αν ναι, υπάρχει αυτή η τυπική μεταφορά τη νομοθεσία, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το πρόβλημα έχει επιληθεί. Okay. Äh, next is... Ευχαριστώ, κύριος Πιέχα. Σας ευχαριστώ. Όπως είπε και ο προλαλής σας, πρόκειται για μία πάρα πολύ σοβαρή έκθεση, αλλά πρέπει να πω ότι πραγματικά είναι απογοητευτικά τα συμπεράσματα, διότι εμείς θα θέλαμε να γίνει κάτι ώστε να αποτραπεί πουν όλα αυτά τα παραποιημένα, τα πλαστά φάρμακα που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάποια στοιχεία για να δούμε ποιες είναι οι ποινικέ κυρώσεις που θα μπορούσαν να επιβληθούν. Αλλά δεν ξέρω ποια είναι η κλίμακα παραποίησης. Δεν ξέρω τίποτε καινούριο σε σχέση με αυτά που ήξερα ε, στο παρελθόν. Και βεβαίως μέσω διαδικτύου ξέρουμε ότι κυκλοφορούν πάρα πολλά πλαστά φάρμακα. Η Επιτροπή μπορεί να μας κάνει κάποιες ε, υποδείξεις για να δούμε πώς θα μπορέσουν τα ε, ηλεκτρονική, ηλεκτρονική διεύλη διανομής τέτοιου είδους παραποιημένων φαρμάκων να ε, υπακούσουν σε κάποιους κανόνες. Επίσης υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα, σκευάσματα, φαρμακευτικά, ε, προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε συμπληρώματα διατροφής. με διά, κυκλοφορούν διάφορα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται από άτομα τα οποία θέλουν να αλλάξουν τη διατροφή τους ή γυμνάζονται και ξέρουμε ότι πολύ συχνά περιέχουν διάφορα παραποιημένα συστατικά. Δεν ξέρουμε πολλά πράγματα για το θέμα αυτό. Επίσης, θα πρέπει να μιλήσουμε και για τα καλλιντικά, διότι εδώ δεν αναφέρονται τα καλλιντικά. Θα πρέπει όμως, διότι όντως τα καλλιντικά περιέχουν διάφορες ουσίες φαρμακευτικές οι οποίες θα μπορούσαν να παραποιηθούν και να ε, οδηγήσουν σε σοβαρέ νοσήματα. Καρκίνο, Φερρυπίν. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Η κυρία Κάντεμπαχ τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Πίτερ Λίζε, γιατί από τη μία έχουμε το θέμα της ανεκνευσιμότητας και έχουμε το θέμα τον κυρώσεων. Αυτό τόνισε. Τα δεδομένα έχουν να κάνουν κυρίως με το εμπόριο, αλλά αυτό που θα με ενδιαφέρει να ξέρω είναι το εξή. Ε. Όταν ξεκίνανε τελικά δικαστικές διαδικασίες, τα κράτη-μέλη προσπαθούν να στραφούν, να κοιτάξουν και πέρα από το συγκεκριμένο έμπορο που προώθησε τα φάρμακα αυτά, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε και που παράγονται τα φάρμακα αυτά, να διαπιστώσουμε από ποιες πηγές προέρχονται. Εκεί λοιπόν αυτό ερευνάτε, Υπάρχουν τέτοιε δικαστικέ διαδικασίε, συμφωνίε, ενδεχομένω και με τρίτα κράτη-μέλη. με άλλε χώρε οι οποίε ενδεχομένω να συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην παραποίηση των ε, φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων. Μάλιστα, λέει Πρόεδρο, δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει να πάρει το λόγο. Να δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δέκα λεπτά έχετε για να απαντήσετε. Okay. Συγγνώμη, η κυρία Καβεθών είχε ζητήσει το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Όντως, στο ίντερνετ και στα ηλεκτρονικά δίκτυα διανέμονται όλα αυτά τα παραποιημένα φάρμακα. Σε εθνικό επίπεδο και η επιβολή κυρώσεων κάτι έκαναν ώστε να περιοριστεί αυτό το εμπόριο αν θέλετε. Αλλά δεδομένου ότι δεν υπάρχουν στο ίντερνετ όρια τι είδου ε, πληροφορίες μπορούμε να έχουμε σε επίπεδο κρατών μελών για να ξέρουμε εάν ε, κάποιες πληροφορίες οι οποίες αποκαλύπτονται σε μια χώρα μπορούν ε, να είναι πληροφορίε από τις οποίες θα υποφεληθούν και άλλοι. Δεν ξέρω αν υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμό. Υπάρχει συγκεκριμένο επίση κατάλογος των εν λόγω πλαστών φαρμάκων ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για να δω. Κανένας άλλος ζητά το λόγο. Η Επιτροπή λοιπόν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Αρχίζοντας, θα ήθελα να πω το εξής, όσον αφορά την κλίμακα του προβλήματος. ένα από, με, από 10.000 σκευάσματα είναι παραποιημένα. 3% λοιπόν των σκευασμάτων όντως είναι παράνομα. Είναι σημαντικό το πρόβλημα. Η έκθεση που εγκρίναμε, που παρουσιάστηκε σήμερα εδώ, περιορίζεται στο να δώσει μια γενική επισκόπηση στο πώς έχουν εφαρμόσει τις κυρώσεις στα κράτη-μέλη και να γίνει εκτίμησή τους, αξιολόγησή τους. Περί αυτού πρόκειται στην έκθεση. Αλλά θα ήθελα να αναφερθώ και σε διάφορα άλλα μέτρα τα οποία λαμβάνουμε ώστε να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα και σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη, βεβαίως. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε ένα σύστημα ε, γνησιότητας των φαρμάκων με κάποια χαρακτηριστικά ειδικά. Με το, αυτό το σύστημα θα εφαρμοστεί από το Φεβρουάριο 2019. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συνεργαζόμαστε εκ του σύνεγγες με τα κράτη-μέλη και με την φαρμακοβιομηχανία ώστε να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμογή πλήρως το σύστημα αυτό σε ένα χρόνο. Πρόκειται λοιπόν για ένα σημαντικό εργαλείο που θα μας βοηθήσει στην ανιχνεσιμότητα των πλαστών φαρμάτων. φαρμάκων. Θα συνεχίσουμε με τα κράτη-μέλη να κάνουμε ελέγχους ώστε πραγματικά να εφαρμοστούν πραγματικές κυρώσεις και αποτελεσματικές τα κράτη-μέλη. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να μπορούν να ελέγχουν κατά πόσο σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία και ε, επιβάλλονται κυρώσεις. Βεβαίως ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, μεγάλες ε, διαφορές μεταξύ κρατών μελών και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον έλεγχο. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι ο φαρμακοβιομηχανία είναι υπεύθυνη, αν θέλετε, για το τελικό προϊόν το οποίο διατίθεται στην αγορά. Και όταν αγοράζονται, ε, ακόμη και όταν αγοράζει κάποιες από τις ουσίες που χρησιμοποιείται σε τρίτες χώρες. Δεν υπάρχει ε, βάση δεδομένων σε κοινοτικό επίπεδο για τον έλεγχο των ενδελεχή, αλλά είμαστε σε συνεχείς συνεδριάσεις και συζήτηση με τα κράτη-μέλη για να παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Ποια άλλη δράση αναλάβαμε για τις ε, πωλήσει μέσω διαδικτύου και ξέρουμε ότι έχουν γίνει διάφορες ερωτήσεις από τους συναδέλφους σας. Δεν έχουμε ε, συγκεκριμένους αριθμούς για το πρόβλημα αυτό. Είναι και πάλι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν μετρήσεις, δεδομένου ότι πρόκειται για μια παράνομη εμπορική δραστηριότητα. Όντως όμως είναι ένα θέμα σημαντικό. Ξέρουμε ότι κάποιοι καταναλωτές, χωρίς να το γνωρίζουν, αγοράζουν τέτοιου είδους σκευάσματα το ίντερνετ. Και έχουμε ένα, αναπτύξει ένα λογότυπο το οποίο πρέπει να φέρουν όλα τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, αν θέλετε, ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι αγοράζουν φάρμακα που δεν είναι πλαστά. Τώρα, για να αυξήσουν ε, την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το λογότυπο αυτό, έχουμε φτιάξει έναν ε, ειδικό οδηγό, τον οποίο έχουμε στείλει, ώστε να μπορέσει να υπάρξει άμεση ευαισθητοποίηση, συνειδητοποίηση και να γνωρίζουν οι καταναλωτές ότι τα σκευάσματα τα οποία αγοράζουν μέσω διαδικτύου είναι νόμιμα. Διότι θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι ίδιοι κανόνες ισχύουν εάν πάτε στο φαρμακείο τη γειτονιά αγοράσετε ένα φάρμακο ή αν το αγοράζετε μέσω ίντερνετ. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπουμε κάποια συμπληρωματική δραστηριότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τι εκστρατείε ενημέρωση, αλλά ε, ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ε, εργαλεία που έχουμε θέσει σε, ε, στη διάθεσή τους και να τα προσαρμόσουν στη κάθε εθνική κατάσταση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μάλλον τελειώσαμε. Ε, εξαντλήθηκε η μερίσια διάταξη και εγώ μαζί. Λοιπόν, θα τα πούμε το απόγευμα στις 2.30. 2.30. Γεια σας. Στις 2.30 αρχίζουμε. Λοιπόν, γεια σας.